Okay, so. Μάλιστα. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης, Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ. Είναι η πιο προηγμένη συμφωνία με ε, τις χώρες αυτές. Ο κύριος Λάμστορφ είναι εισηγητής, θα του δώσω αμέσω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μισό λεπτάκι να κλείσω το κινητό. Μπορείτε να βάλετε ακουστικά, συνάδελφοι. Το κλείσα. Αυτή η έκθεση είναι μια έκθεση που θα ε, θα βοηθήσει το Κοινοβούλιο να αποφασίσει τη θέση του. Ο στόχος της συμφωνίας είναι η ενίσχυση των ε, εταίρων μας από τη μία και από την άλλη του εμπορίου με τις χώρες ΑΚΕ, ε, το οποίο τα τελευταία χρόνια δεν είχε την επιθυμητή αύξηση. Πρέπει να εξετάσουμε τη συμβατότητα των εμπορικών μας σχέσεων με τις χώρες ΑΚΕ. Να σας υπενθυμίσω ότι η μεταβατική περίοδος αρχικά ε, έλεγε το 2007, σχεδόν 10 χρόνια πριν. Από τότε είχαμε ε, την ελεύθερη πρόσβαση ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα τέτοιο κατασκεύασμα το οποίο χρησιμοποίησαμε ως μεταβατική λύση. Αυτό που θεωρώ πολύ σημαντικό στην συζήτηση είναι ότι οι χώρες εταίροι μας είναι, ε, βρίσκονται ιονοί υποπίεση και δεν μπορούν να αποφασίσουν ελεύθερα. Μπορώ να δω και να κατανοήσω τους λόγους. Οι εταίροι μας θα έπρεπε να έχουν την δυνατότητα να ε, ταχθούν υπέρ ή κατά μιας τέτοιας συμφωνίας. Οι διαπραγματεύσεις άρχισαν με 7 ε, χώρες, όμως η Αγκόλα αποφάσισε να αποχωρήσει αργότερα, διότι σύμφωνα με εκείνους η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούσε να τους φορέσει στενό κορσέρ. Γι' αυτό λοιπόν τώρα έχουν μείνει έξι χώρες. Δεν συμπεριλαμβάνεται η Αγκόλα. Ε, τώρα, επί του περιεχομένου, πρόκειται καταρχάς για αγαθά και προϊόντα τα οποία ε, έχουν ε, θετική προτιμησιακή αντιμετώπιση. Αυτή η συμφωνία είναι δηλαδή προς το συμφέρον των ε, χωρών εταίρων μας. Υπάρχουν πάρα πολλές ρήτρες διασφάλισης για ε, πολλούς κλάδους, ε, βιομηχανικούς και για συγκεκριμένα προϊόντα, τα οποία παράγονται από λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Είναι βέβαια εκτός από την εμπορική συμφωνία βασικό και ένα άλλο θέμα της περιφερειακής καταγωγής έχω κάποια, έχω, να, έχω κάποια πράγματα στο σπίτι μου, πούμε, που είναι από την Νότια Αφρική και, το, και εάν ισχύει, τεθεί σε ισχύ αυτή η συμφωνία θα προστατεύονται. Επίσης, μείωση των δασμών. Αυτό αφορά ορισμένα αλλιευτικά ε, προϊόντα. Για εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτές ε, οι χώρες ε, εταίροι θα ε, μπορούν από εδώ και μπρος να έχουν, να λαμβάνουν επιδοτήσεις για κάποια αγροτικά προϊόντα. Τώρα, ο τομέας των υπηρεσιών και της, των κρατικών συμβάσεων και της πνευματικής ιδιοκτησίας έχει ακόμα πολλά ε, που πρέπει να γίνουν. Θα χρειαστεί πολλή συζήτηση και στο μέλλον. Αλλά κάτι πολύ σημαντικό είναι η ε, ανάπτυξη και το εμπόριο. Αυτός ο τομέας έχει μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης, πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε, να ε, προωθήσουμε και να στηρίξουμε την ανάπτυξη. Ε, σε πρώτο στάδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ένα ψήφισμά του ζήτησε και μάλλον κατέστησε σαφές ότι το θεωρεί ως προτεραιότητα, όμως μια τέτοια συμφωνία η οποία αφορά εμπόριο αγαθών δεν μπορεί παρά να είναι μέλος μιας μεγαλύτερης, ευρύτερης στρατηγικής. Με αυτήν εδώ τη συμφωνία δεν θα αλλάξουμε δεν θα αλλάξουμε κατεύθυνση στο εμπόριο με αυτές τις χώρες, αλλά πρέπει να το θεωρήσουμε ως ένα ακόμα συστατικό στοιχείο μιας ευρύτερης πολιτικής. Ε, πρέπει να συνδεθεί με το ε, τα Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ανάπτυξη, πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε και αυτό ε, πρέπει να συμπεριληφθεί. Τώρα, κάτι που έχουμε συζητήσει διεξοδικά εδώ και με τους κοιόδης συζητητές, είναι το πώς θα συνοδεύσουμε, με τι θα συνοδεύσουμε την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Ο κύριος Σούστερ και η κυρία Κέρτον Τάρλινγκ ε, γνωρίζουν για αυτά τα θέματα. Μιλήσαμε για εφαρμογή το αργότερο σε πέντε χρόνια και επανεξέταση της συμφωνίας μετά από πέντε χρόνια. Ίσως αυτή θα είναι μια δουλειά του επόμενου κοινοβουλίου, βέβαια, ε, και αναφέρομαι στην συνολική εξέταση της συμφωνίας. Αναφέρεται στο σχέδιο έκθεσης τακτική, τακτικός έλεγχος. Ε, υπάρχουν και οι αντίστοιχες δομές τις οποίες, οι οποίες θα το βοηθήσουν. Φυσικά πρέπει να βελτιώσουμε το κείμενο. Αυτό που έχουμε προσπαθήσει στο ψήφισμα είναι να είμαστε εμείς ε, η ΙΝΤΑ η αρμόδια επιτροπή. Το άρθρο 4 της συμφωνίας βέβαια αφήνει αρκετό περιθώριο ελιγμών για να δημιουργηθούν νέες δομές. Μετά από συνομιλίες με τους ευρωβουλευτές, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τους εταίρους μας από τις χώρες αυτές και με βουλευτές από τα κοινοβούλια των χωρών αυτών. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα ε, να δημιουργηθούν διάφοροι μηχανισμοί επιτήρησης σε συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια. Μπορούμε δηλαδή να δημιουργήσουμε και κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες σε περίπτωση που συναντήσουμε δυσκολίες στην εφαρμογή της συμφωνίας. Τώρα σε γενικές γραμμές θα έλεγα η συμφωνία είναι αρκετά καλή ε, παρότι μας ήρθε 9 χρόνια μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία. Υπάρχει ακόμα δουλειά που πρέπει να γίνει ιδιαίτερα στην, στο μηχανισμό παρακολούθησης, αλλά πιστεύω ότι όλα θα γίνουν στον, στην ώρα τους. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στους κοιόδης εισηγητές, πρώτα με τον κύριο Μάτο από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την έκθεση και μετά να σας πω πως το να συνοψίσουμε σε ένα λεπτό τα αποτελέσματα 10 ετών διαπραγματεύσεων μου φαίνεται λίγο φτωχό. Αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ και να σας πω ποια είναι τα θετικά σημεία της συμφωνίας. Το έκανε βέβαια και ο συγητή με εξαιρετικό τρόπο. Είναι καλή συμφωνία και απαραίτητη συμφωνία, με δύο λόγια. Έτσι είναι τα πράγματα. Και πιστεύω πως η συμφωνία αυτή κλείνει και μία περίοδο νομικής αβεβαιότητας, κάτι το οποίο ήταν απαραίτητο. Γιατί ναι, τώρα πια έχουμε το διμερές και περιφερειακό νομικό πλαίσιο με ένα πλαίσιο που συμβαδίζει και συμμορφώνεται με τους κανόνες του ΠΟΕ, κάτι το οποίο ήταν απολύτως απαραίτητο. Δεν πρόκειται να μιλήσω για τις διάφορες διατάξεις και τις ρήτρε, απλώς θα τονίσω πως έχουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη που δείχνει πως και τα δύο μέρη ανησυχούν ε, για το θέμα αυτό και να ε, υπογραμμίσω την περιφερειακή διάσταση αυτής της ε, συμφωνίας που εναρμονίζεται με την Τελωνιακή Ένωση και που ενδεχομένως θα είναι ένα συμπληρωματικό στοιχείο που θα προσφέρει κάτι σε αυτήν την Ένωση. Και επειδή εγώ είμαι από τα Κανάρια νησιά που είναι πολύ περιφερειακή περιοχή και πάντα η καρδιά μου το αισθάνεται, πιστεύω πως επειδή ακριβώς αποκλείσαμε την βιομηχανία ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο, κάναμε κάτι πάρα πολύ καλό, γιατί έτσι διατηρούμε την, ελληνική, την ευρωπαϊκή ε, βιομηχανία. Ξέρω ότι για τους Γάλλους στην περιφέρεια υπάρχει πρόβλημα, αλλά καταλαβαίνετε πως αυτή τη στιγμή που το, οι ζάχαρης ε, πρόκειται να εξαλειφθούν, νομίζω πως αυτό που κάναμε είναι πάρα πολύ σωστό και μαζί με τα υπόλοιπα που τονίσαμε ήταν καλό και αυτό. Χαίρομαι που έχει υπογραφεί και η ομάδα η δική μας θα στηρίξει και θα εγκρίνει απόλυτα αυτή τη συμφωνία. Έχω την εντύπωση ότι ε, μαζί με την ε, Μαρία Αρένα πρέπει ε, να δούμε και τι γίνεται με όλη την ε, συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΚΕ. Εγώ προσωπικά δεν έχω ακούσει από κανέναν ε, βουλευτή χωρών και να λέει πως είναι ευχαριστημένος από αυτή τη συμφωνία. Αυτά έτσι προκατακτικά. Εγώ πιστεύω πως πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη τις αντιρρήσεις και τις ανησυχίες και τους ε, δισταγμούς που έχουν οι εταίροι μας, διότι πέρα από τις ευκαιρίες που παρουσιάζει, ε, περιέχει και πολλούς κινδύνους. Ναι, μεν θα στηριχθούν οι οικονομίες των χωρών αυτών, όμως ε, δεν συμπεριλαμβάνονται όλες οι χώρες στη συμφωνία αυτή. Και αυτό πιστεύω πως δεν είναι θετικό. Τώρα, αυτή η ρήτρα που ανέφερε ο κύριος Λάμστορφ είναι κάτι που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Θα προστατευτεί ε, η βιομηχανία, ιδιαίτερα οι νέες επιχειρήσεις, όμως πρέπει να δούμε πότε θα εφαρμόζεται και ε, αυτή η ρήτρα εφόσον παρατηρηθούν δυσλειτουργίες. Επίσης, να σας πω ότι αυτή η συμφωνία είναι, ε, δεν είναι κάτι το υποχρεωτικό, ιδιαίτερα με την Νότια Αφρική, η οποία είναι μια κυρίαρχη οικονομία στην περιοχή. Και ας μην ξεχνάμε ότι ως κυρίαρχη οικονομία ασκεί και πίεση στις πιο δύναμες ε, χώρες οικονομικά της περιοχής. Ε, τα πράγματα λοιπόν δεν είναι και τελείως ε, εθελοντικά. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ναι, μεν πρέπει να ασκήσει πίεση, αλλά αυτό μπορεί να το κάνει μόνο μέχρι τι αρχέ Οκτωβρίου και το γεγονό ότι καθυστερήσαμε 10 χρόνια μέχρι να φτάσουμε σε αυτό εδώ το σημείο είναι κάτι που ε, θεωρώ κατανοητό μετά από όλα που έχουν γίνει. όμω από εδώ και μπρο οι καθυστερήσει είναι αδικαιολόγητε. Εάν καθυστερήσει η επικύρωση τη Συμφωνία πάνω από τρει μήνε υπάρχουν κυρώσει. Και πιστεύω πως αυτή η πίεση είναι δυσανάλογα μεγάλη σε αυτό το στάδιο. Επίσης πρέπει να είμαστε σε θέση να δεχτούμε και, ένα, ε, και μια αρνητική απόφαση. Αν το Κοινοβούλιο δηλαδή αποφασίσει να καταψηφίσει, αυτό πρέπει να το ε, δεχτούμε. Τώρα, να τονίσω και κάτι άλλο. Ο κύριος Λάμστορφ το είπε νομίζω κιόλα, η εφαρμογή και η παρακολούθηση. Εάν θέλουμε να έχουμε θετική τα αποτελέσματα από την, εφαρμογή, από την συμφωνία, πρέπει να παρακολουθούμε την εφαρμογή της για να μπορούμε να ελέγξουμε το κάθε και να δούμε τι γίνεται, για παράδειγμα, για τη βιώσιμη ανάπτυξη, πώς αυτή η συμφωνία ευνοεί ή βλάπτει τη βιώσιμη ανάπτυξη και γι' αυτό θα ήθελα να συμφωνήσω με τον κύριο Λάμστορφ και να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ε, αφήσει να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο που έχουμε μέχρι την ε, κύρωση της, της συμφωνίας για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το περιεχόμενό της, να δούμε πόσο μπορούμε να ενσωματώσουμε τις αξίες μας στο κείμενο και πώς μπορούμε να αποκομίσουμε ωφέλη για την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κέμπελ λείπει νομίζω ή όχι. Ποιος έχει σειρά. Ευχαριστώ κύριος Υπουργός ε, δεν είναι εδώ για προφανείς ε, λόγους. Θα ήθελα λοιπόν απλώς ε, να σας αναγνώσω την γνώμη του ως Γιώδους. Χαιρετίζει τη συμφωνία που ενισχύει τις σχέσεις με τις χώρες της ΚΑΜΑ σε ένα εύρωστο πλαίσιο ε, που συνάδει με τους κανόνες ε, ΠΟΕ, γιατί προηγουμένως αυτό δεν ίσχυε. Ε, χαιρετίζουμε λοιπόν τις συστάσεις του εισηγητή, το Ευρωκοινοβούλιο να συνενέσει. Για το ECR η πιο σημαντική πτυχή της συμφωνίας είναι ότι οι πτυχές ανάπτυξη του εμπορίου θα εφαρμόζονται πλήρως, ώστε αυτέ οι χώρε να εξακολουθούν να υποφελούνται τη ε, άνευ δασμών πρόσβαση στην ε, ευρωπαϊκή αγορά. Εάν αξιοποιηθούν αυτέ οι δυνατότητε, πρέπει επίση η Ευρωπαϊκή Ένωση να του βοηθήσει με ε, εμπορικά συστήματα για να αναπτύξουν τι ικανότητε του και έτσι καλύτερα να μπορέσουν να ενσωματωθούν στι παγκόσμιες αγορέ και αλυσίδε αξιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Φορέντσα από το πλευρά Γκουέ δεν είναι εδώ όμω, ο κύριο Σόλτ. Ε, <clears throat> Εγώ είμαι ο Σκιώδη. Α, συγγνώμη, δεν έχει, τα έχουμε σημειώσει σωστά. Γιατί είμαι και εισηγητή ε, για την ε, κοινότητα για την Ανατολική Αφρική. Συμφωνώ πλήρω με τα όσα είπε ο κ. Σούλστερ για το περιεχόμενο της συμφωνία. Όμως, επιπροσθέτως, ένα τεχνικό, διαδικαστικό, θεσμικό ζήτημα προς την Επιτροπή. Την περασμένη φορά που υπήρξε ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό, δεν υπήρξε καμία ενημέρωση ότι θα υπάρξει συνεδρίαση της ε, ομάδας πρόσβασης ε, στην αγορά και ότι θα υπάρξει τέτοια ανάλυση τη κατάσταση ό,τι αφορά αυτέ τι έξι χώρε. Επομένω, θέτω αρχικά το ερώτημα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο εισηγητή εν μέρη μας έχει ενημερώσει. Υπάρχουν ενδείξει ότι κάποια από τι χώρε τη Ανατολική ή Μεσηβρινή Αφρική δεν προτίθενται να κυρώσουν την ε, ΣΟΕΣ αυτή. Γιατί λοιπόν αυξάνεται τι πιέσει προ αυτέ τι χώρε. υπό την απειλή μάλιστα ε, άρσης ε, των, ε, της προτιμησιακής μεταχείρισης. Την 1η Ιουνίου μόλις ε, το Συμβούλιο αποφάσισε να κυρώσει ε, την απόφαση αυτή. Δεν έχει αποφασίσει λοιπόν να υπογράψει. Γιατί λοιπόν αυξάνονται αυτές οι πιέσεις εάν δεν κυρωθούν συμφωνίες από τις ε, χώρες ε, αυτές. Θα πρέπει εκεί να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο μέχρι τον Οκτώβριο του 2016. Επομένως ε, δεν κατανοώ γιατί δημιουργείται αυτό το ζήτημα και νομίζω ότι αυτό είπε και ο κ. Σούλουστερ μετά την συνάντηση με τις χώρες ΑΚΕ. και μετά τη συνάντηση ΠΟΕ. Ακόμα και ως εκπρόσωπος ε, του Γερμανικού Κοινοβουλίου από πλευράς ΕΛΚ. Μάλιστα, ο ίδιος είχε αναφέρει με, σημαντικό, με μεγάλο προβληματισμό ότι ήταν ε, ιδιαίτερα επιταχυμένη διαδικασία και δεν ε, αυξάνεται η εμπιστοσύνη. Και δεν χρησιμοποιούμε το εμπόριο ως εργαλείο ανάπτυξης κάνουμε το αντίθετο. Αυτό είναι το ερώτημά μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αν μπορείτε και πάλι να μας εξηγήσετε την νομική βάση για τον οδικό χάρτη που έχετε καταρτήσει σε ό,τι φορά την κύρωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Από πλευρά Πρασίνων. Φυσικά και Έχουμε εδώ, αλλά μάλλον φαντάζομαι εδώ θα την αντικαταστήσετε. Νομίζω ότι και επισήμω το έχουμε αλλάξει αυτό πριν από καιρό. Τέλο πάντων, δεν πειράζει. Δύο ερωτήματα μόνο, γιατί τα περισσότερα έχουν ήδη υποθεί από του κυρίου Σούσλε και Σόλτ. Προς τι τόσο βιασύνη. όντω. Ο εισηγητή ε, παρουσίασε πολύ σωστά την κατάσταση. όντω ήταν μακροσκελή η διαδικασία, υπογράφει, υπεγράφει όμως στι 10 Ιουνίου. Θα πρέπει να εφαρμοστεί τον Οκτώβριο. Γιατί ξαφνικά λοιπόν βιαζόμαστε τόσο και, και γιατί είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο. Ιδάλω αυτέ οι χώρε θα χάσουν την πρόσβαση στην αγορά του. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί υπάρχει τέτοια βιασύνη. Και το δεύτερο ερώτημα. Υπάρχει τώρα συζήτηση ε, στην Αφρική ε, για ελεύθερη ζώνη συναλλαγών ε, στην Ήπειρο. Εμείς έχουμε και αυτό το ΙΠΑΣ, πώς, μάλλον έχουμε τις περιφερειακές ΣΟΕΣ και πώς θα διαβεβαιώσουμε ότι δεν θα υπάρξει αρνητική αλληλεπίδρυση. Ευχαριστώ, Μαρία. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε τον εισηγητή και τον συνεισηγητή με μεγάλη προσοχή διάβασα την ε, γνωμοδότηση του κ. Λαμσδόρφη και συμφωνώ με τα όσα είπε ο Ζωακίν. Ε, τώρα έχουμε μία ιδιαίτερη τέτοια συμφωνία ΣΟΕΣ γιατί εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ε, πλαίσιο της συμφωνίας Κοτονού. Και εδώ έχουμε και ψήφισμα στο Κοινοβούλιο με το οποίο θετήσαμε τέσσερις βασικές αρχές που νομίζω ότι δεν τηρούνται στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας. Πρώτη αρχή οφείλουμε να μεριμνήσουμε ώστε να μην στείλουμε προϊόντα στην Ευρώπη που λαμβάνουν επιδοτήσεις σε σχέση με τα αφρικανικά προϊόντα. Ξέρουμε ότι υπάρχει ε, προτιμησιακό καθεστώς ε, για απέναντι στην Αφρική που τελικά οδηγεί στην στήριξη ορισμένων ε, παραγωγών, ιδίως ότι φάτε γεωργικά προϊόντα. Και όντως εδώ τα γεωργικά προϊόντα είναι ευαίσθητα προϊόντα και θα επανέλθω σε αυτό για τι αφρικανικέ χώρε, όμω έχουμε τη δυνατότητα εξαγωγή ε, συγγνώμη, γεωργικών ε, προϊόντων ε, όπου υπάρχει dumping σε σχέση με τη δική μα πολιτική. Μιλούμε για την Κίνα για το dumping, αλλά για εμά δεν λέμε στην Ευρώπη όταν υπάρχει dumping για τα δικά μα προϊόντα που και τα στέλνουμε τελικά στην Αφρική. Εδώ είναι η πρώτη αρχή που ήδη παρουσιάζει προβλήματα για τα ευαίσθητα προϊόντα. Δεύτερη αρχή, ευελιξία ως προς τα, ε, τα φρολικά σύνορα. Ξέρετε ότι σε ορισμένε συμφωνίε άλλε χώρε δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα να παίξουν λίγο με αυτά τα ζητήματα, τα φορολογικά. Ένα κέντρο Αφρικανικών Επιστημών ε, Μελετών δείχνει ότι οι Αφρικανικέ χώρε χάνουν 3,5 δι έσοδα ακριβώ λόγω τη κατάργηση αυτή τη δυνατότητα με τα φορολογικά του σύνορα. Όμω είναι ένα από του τρόπου που έχουν να προστατεύσουν τμήμα και τη τοπική του οικονομία. Με αυτόν τον τρόπο πράγματι υπάρχει μια ρήτρα που επιτρέπει την προστασία της τοπικής οικονομίας, το infant clause, όμως είναι τόσο δύσκολο να εφαρμοστεί αυτή η ρήτρα που η τοπική οικονομία ουσιαστικά αργοπεθαίνει πριν καν ε, τεθεί σε ισχύ αυτή η ρήτρα. Γι' αυτό και ο κύριος ε, Λάμστορφ το λέει στην έκθεσή του, ότι πρέπει να ε, συγκεκριμένη και υποχρεωτική παρακολούθηση, ούτω ώστε ακριβώ να εφαρμόσετε σωστά αυτή η ρήτρα. Τρίτη αρχή, σε ό,τι αφορά τους κανόνες ε, προέλευσης και την ε, ελαστικοποίησή τους. Ε, υπάρχει αυτή η πτυχή, όμως όταν θα πρέπει να υπάρξει εξαγωγή βόλιου κρέατος από την Αμήμπια θα έχουν πολύ μεγαλύτερη δυσκολία να το πράξουν σε σχέση με τους Καναδούς, για παράδειγμα, στη ΣΕΤΑ. Γιατί και εκεί η ΣΕΤΑ θα καταστήσει πολύ δύσκολη και την συμφωνία αυτή με τις χώρες ΚΑΜΑ. Και τέλος, το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης, πράγματι υπάρχει το κεφάλαιο βιώσιμης ανάπτυξης, μοναδική συμφωνία σήμερα με την Αφρική που προβλέπει τέτοιο κεφάλαιο. Δυστυχώς όμως αυτό το κεφάλαιο δεν έχει καμία υποχρεωτική ρήτρα. Όμως ε, νομίζω ότι η Ευρώπη καλό θα τη κάνει να είναι πιο ε, ειλικρινής ως προς την τη. της. Να λέμε λοιπόν ότι κερδίζει πολλά η Ευρώπη από αυτή τη συμφωνία. Απελευθέρωση στο 86% της αφρικανικής αγοράς, που δεν είναι αυτό που ζητάει ο ΠΟΕ. Πάμε λοιπόν πιο μακριά από αυτό που ζητάει ο ΠΟΕ ε, ως προς την απελευθέρωση. Συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων γεωργικών και αλευτικών προϊόντων. Δεύτερον, ο κατάλογος των ευαίσθητων αυτών προϊόντων. Εγώ θα ήθελα να είναι αθρηστικός. Σήμερα υπάρχει συμφωνία που λέμε ότι υπάρχει κατάλογος τέτοιος για την Αφρική, αλλά δεν είναι τα ίδια τα ευαίσθητα προϊόντα για την Αμίμπια και τη Σουαζιλάνδη. Αυτό τι σημαίνει, ότι ένα ευαίσθητο προϊόν δεν πρέπει δηλαδή να μπει στην επικράτεια της Ναμίμπιας, θα μπει όμως από την Νότια Αφρική. Και καθώ έχουν ε, εσωτερική ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, ένα ευαίσθητο προϊόν που δεν θα μπορούσε να έχει μπει στην Αμίμπια, μπαίνει από την Νότια Αφρική και φτάνει τελικά μέσω Νότια Αφρική στην Αμίμπια. Είναι σαν να λέγαμε ότι υπάρχει ευαίσθητο προϊόν στο Βέλγιο που δεν είναι ευαίσθητο προϊόν στη Γερμανία. Εντάξει, θα πάει από τη Γερμανία και θα μπει στην εσωτερική αγορά και έτσι θα απολυθεί τελικά και στο Βέλγιο. Αυτό κάνουμε ουσιαστικά. Ουσιαστικά καταστρέφουμε την εσωτερική του ε, δομή. Εγώ θα προτιμούσα λοιπόν έναν ανθρεστικό κατάλογο ευαίσθητων προϊόντων που δεν θα επέτρεπαν την εισαγωγή τους ε, από την πίσω πόρτα. Ε, επίσης, η Ευρώπη κερδίζει και σε ό,τι αφορά τα λοιπάσματα. Ε, διασφαλίζουμε την παρουσία των λοιπασμάτων που παρασκευάζονται μάλιστα στην Ευρώπη στην Αφρική. Κερδίζουμε λοιπόν για να στηρίξουμε υπερεντατική γεωργία σε χώρες όπου έχει τεράστια αλληψιδρία και αυτό θα πλήξει τον τοπικό πληθυσμό. Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν. Υπάρχει ε, ανά πέντε έτη ρήτρα αναθεώρηση. Θα σα πει και ο εισηγητή ότι σε αυτή τη ρήτρα αναθεώρηση δεν έχουμε μόνο τη βελτίωση σε σχέση με τα όσα δεν λειτουργούν καλά, όμως ε, επεκτείνεται η συμφωνία στις υπηρεσίες, ε, στις ε, δημόσιες συμβάσεις, στα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησίας. Υπάρχει στην έκθεσή σας, αλλά όχι στην αιτιολόγηση. Ποιος επωφελείται από όλα αυτά. Σίγουρα όχι οι Αφρικανοί. Ξέρετε πολλούς Αφρικανούς που θα, θα εφτάσουν στην ευρωπαϊκή αγορά, στις ε, δημόσιες συμβάσεις, δεν νομίζω. Αντιθέτως για την Ευρώπη θα την ευνοήσει. Και βέβαια, και πολύ σημαντικό, δεν υπάρχει καμία αποζημίωση ό,τι αφορά τα μέσα ανάπτυξης. Μηδέν, απόλυτο μηδέν. Ε, Πήγατε στην ε, Ναμίβια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξαφνικά, βεβαίω, επειδή ήταν ε, να υπογράψετε, όλοι ήταν πλήρω ευχαριστημένοι. Είπατε ότι χρειάζεται ένα δεύτερο πρόγραμμα ΦΕΔ, χωρίς ε, κανένα, λοιπόν, χωρί καμία επιπρόσθετη χρηματοδότηση. Επομένω, θα πρέπει να πληρώσουν εκείνοι το κόστο ε, προσαρμογής. Δηλαδή, τελικά, είναι απίστευτο. Δεν θα στοιχήσει τίποτα στην Ευρώπη. Όμω εκεί που υπάρχουν ζητήματα προσαρμογή. Ποιο θα τα καλύψει αυτό το, το κόστο. Δεν το θεωρώ σωστό αυτό. Μπορούμε να στηρίξουμε μια τέτοια συμφωνία αν αποδεχθούμε ότι θα δώσει περισσότερα πλεονεκτήματα στην Ευρώπη παρά στην Αφρική, να το παραδεχθούμε δηλαδή, και δεύτερον, τις ζημίες αυτές να τις καλύπτουμε που, δημιουργούμε στην Αφρική. Να τις καλύψουμε, να μην είμαστε υποκριτές σε αυτή την έκθεση, σε αυτή τη συμφωνία, συγγνώμη. Και θα ήθελα οι ρήτρε αυτές, οι συνοδευτικές, ε, ε, όντω να τεθούν σε λειτουργία. Όπω είπε πολύ σωστά και ο συγγετή, να αναφερθώ κι εγώ σε ό,τι αφορά την, ε, το σεβασμό προ τα κοινοβούλια. Είναι απίστευτο. Θα τεθεί σε ισχύ συμφωνία χωρί να περάσει. Η κυρία Πλούμαν από την Προεδρία του Συμβουλίου χθε είπε «Εγώ δεν είμαι υπεύθυνη για την δημοκρατία στην Αφρική». Ισχύει. Δεν έχουμε εμεί αυτή την ευθύνη. Όμως, το να κάνει κανεί αυτό που κάνατε εσεί, να του βάλετε το μαχαίρι στο λαιμό, ότι Ναμίμπια, Σουαζιλάνδη, Μποτσουάνα, αλλά και υπόλοιπε χώρε, ε, Κένια και άλλε που αντιτίθεται περισσότερο στην ελεύθερη ζώνη συναλλαγών, δεν θα έχουν πρόσβαση στην αγορά εάν δεν κυρώσουν μέχρι την 1η Οκτωβρίου, ενώ δεν υπάρχει καν υπογραφή, δεν θα έχουν δηλαδή καν ένα μήνα να τα συζητήσουν στο κοινοβούλιο του. παρότι δεν έχουμε βρει ούτε έναν βουλευτή στην διακοινοβουλευτική ΑΚΕ. Ούτε έναν δεν βρήκαμε που να γνωρίζει τι συμβαίνει στι διαπραγματεύσει. Κανεί δεν είχε γνώση λοιπόν των διαπραγματεύσεων. Ούτε ένα. Ούτε αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι σωστό. Δεν σεβόμαστε με αυτόν τον τρόπο τι αφρικανικέ δημοκρατίε. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για αυτέ, όντω, αλλά ούτε μπορούμε να, ακριβώ να προβούμε σε αυτή την καταστροφή ε, τη δημοκρατία στην Αφρική. Ευχαριστώ. Να σας πω στα γρήγορα, γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά από τους συναδέλφους και κυρίως από τους ε, σοσιαλιστές. Αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον, αλλά παράλληλα ε, είναι ε, και ντροπή για μας, είναι ότι αυτή η συμφωνία είναι η μη χείριστη. Εντάξει, γιατί δεν είναι δεσμευτικό το περί, περιβιώσιμης ανάπτυξης, γιατί η συμφωνία αυτή είναι πιο ασυμμετρική ασύμμετρη από ό,τι άλλε αντίστοιχε, γιατί προστατεύονται οι γεωγραφικέ ενδείξει, αλλά όχι Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα τα οποία επιμένουν και επειδή και η Μαρία και ο Ιωακήμ ε, επιμένουν, να σας πω πως το πρώτο πρόβλημα για μένα είναι περισσότερο συμφωνία εμπορική παρά αναπτυξιακής βοήθεια Δηλαδή, κάποια προβλήματα δεν τα λαμβάνουμε παρκώς υπόψη. Δηλαδή, τι θα μπορούσε ε, να επιβάλλει ένα καθεστώς κυρώσεων για, ένα, ε, για μια κυβέρνηση που δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν έχουμε κάτι το αυτόματο που ενεργοποιείται. Και ε, εδώ τα συμφέροντα που πριτανεύουν είναι ξεκάθαρα εμπορικά. Ε, έχουμε συναδέλφους που δεν είναι εδώ, όπως ο Ντόμ Ντάρλινγκ που είχε πει πως η διατάξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτή τη συμφωνία είναι ε, λιγότερα από αυτά που έχουμε με την Κολομβία, το Περού ή με τις χώρες της Καραϊβικής. Νομίζω ότι αυτό είναι πρόβλημα. Δεύτερον, ο Γιωακίμ το είπε και θα επανέλθω. Εμείς την περιφερειακή ολοκλήρωση δεν την ευνοούμε με τον τρόπο αυτό, γιατί δίνουμε διαφορετικές παραχωρήσεις ανάλογα με τη χώρα και αυτή τη στιγμή οι δομές ε, που σχεδιάζουμε δεν είναι τόσο επαρκείς όσο υπάρχουσες. Τρίτον, ε, κοινωνία των πολιτών και η εμπλοκή αυτής και των πολιτών. Ξέρω πως για αρκετούς από τους συναδέλφους ε, έγινε μια προσπάθεια από πλευρά του ένα είδο πρωτόκολλο για το θέμα αυτό να ενταχθεί στη συμφωνία, αλλά δεν υπάρχει ακόμα. Και τέταρτον, το είπαν αρκετοί συνάδελφοι και πάλι θα σταθώ σε αυτό. Η πίεση που δεν ζητά να εφαρμόσει από την Κομισιόν ΟΠΟΕ. Είπε προθεσμία 1η ε, Οκτωβρίου του 2016. Ναι, Εντάξει, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή η στάση που ακολουθούμε αξίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, το να υποκύπτουμε σε τέτοιου είδου πολιτικέ πιέσει δεν μα τιμά. Και νομίζω ότι θα πρέπει να βγούμε με το κεφάλι ψηλά, αλλά να βρούμε ποια θα είναι αυτή η λύση που θα μα επιτρέψει. Και έχω αρκετέ συμφωνίε ακόμα για αυτή τη συμφωνία που συζητάμε. Κρίστοφ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Δυσκολεύομαι και εγώ να δω για ποιο λόγο βιαστήκαμε τόσο πολύ, για ποιο λόγο πιεστήκαμε τόσο πολύ, αφού δέκα χρόνια το συζητάμε. Και το περιεχόμενο είναι γνωστό εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν μπορώ καν να μετρήσω πόσες συνεδριάσεις κάναμε σε αυτή την Επιτροπή και σε άλλες Επιτροπές για το θέμα αυτό. Συζητήσαμε το περιεχόμενο, αξιολογήσαμε το περιεχόμενο. Εάν κάποιος επιχειρηματολογούσε και έλεγε πως χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο και να έχουμε ένα πιο λογικό ε, χρονοδιάγραμμα. Θα ήθελα να πει ποιο ακριβώς είναι το λογικό χρονοδιάγραμμα αφού έχουμε χάσει τόσο χρόνο ήδη. Πάντως εδώ η σύγκριση που γίνεται είναι μεταξύ του πώς εμείς αντιμετωπίζουμε και βλέπουμε την Αφρική. Και θα ήθελα να σας δώσω μία άλλη ε, οπτική γωνία σε σχέση με αυτή που παρουσίασαν τώρα οι συνάδελφοι κυρίω. Γνωρίζουμε πως η ανησυχία που εκφράζεται δεν έχει για το πώς θα επηρεάσει η συμφωνία αυτή. Εντάξει, για τις αγορές δεν υπάρχει πρόβλημα και για τους πολίτες μας. Η ανησυχία μας είναι πώς θα επηρεάσει τους Αφρικανούς εμπορικούς μας εταίρους. Το περασμένο Σάββατο, νομίζω, υπεγράφει από μία σειρά νομίμων, δημοκρατικά εκλεγμένων ε, υπουργών ε, εμπορίου από τη Ναμίμπια, από την Νότια Αφρική και άλλα κράτη και αυτή τη στιγμή συζητάμε εάν έκαναν μια σωστή επιλογή, μια λογική επιλογή για να υπογράψουν. Δηλαδή, εάν έκαναν αυτό το οποίο εξυπηρετεί τα συμφέροντα του δικού τους κράτους. Αυτό συζητάμε. Και εγώ Βρίσκω μόνο δύο επιχειρήματα γιατί η Επιτροπή δική μας θα έλεγε όχι σε αυτή την διαπραγμάτευση. Και είναι ότι ή εμείς ξέρουμε τη δουλειά σας καλύτερα από εσάς, κοιτάξαμε το κείμενο και εσείς δεν το έχετε καταλάβει, δεν ξέρετε τι συνέπειες θα έχετε για εσάς, εμείς θα ξέρουμε καλύτερα αυτά τα πράγματα, ή, γιατί μόνο η άλλη είναι η εναλλακτική λύση, είναι ότι λυπάμαι, εσείς οι υπουργοί δεν νομιμοποιήσετε να λάβετε αυτή την απόφαση. Μιλάμε τώρα για μια νεοαπικιοκρατική αντίληψη που είναι θλιβερή. Σε μια ε, στιγμή που η Αφρική βρίσκεται στα πιο αναπτυγμένα της, στα πιο δημοκρατικά της και λέμε εντάξει περισσότερο αναπτυξιακή βοήθεια παρά εμπόριο. Μα συγγνώμη, πέρασαν οι καιροί και η Αφρική πια χρειάζεται εμπόριο, όχι αναπτυξιακή βοήθεια. Άρα λοιπόν εντάξει, μπορείτε να ονειρεύεστε το ποια ήταν η παλιή καιρή και ποιε ήταν οι παλιέ συγκρούσει. Αν έλα να αξιολογήσουμε αυτή την συμφωνία, την αξιολογήσουμε με τη βάση, στη βάση του τι είναι Αφρική σήμερα. Που είναι ε, νομιμοποιημένε δημοκρατικέ ε, κυβερνήσει, οι οποίε γνωρίζουν ε, επαρκώ το τι τι εξυπηρετεί και όχι. Οπότε, αφού αυτοί το ε, υπέγραψαν, εγώ θα το επικυρώσω με χαρά. Ε, ο κύριος Σούλτ έχει το λόγο για μια σύντομη παρατήρηση. Λοιπόν, για να δούμε τα θέματα, τα συνταγματικά που προκύπτουν. Και μπορείτε να μου απαντήσετε, γνωρίζετε να υπάρχει οποιοδήποτε συνταγματικός κανονισμός στις χώρες για τις οποίες συζητάμε που θα τους επέτρεπε να υπογράψουν μια συμφωνία την οποία δεν έχουν συμφωνήσει σε εθνικό επίπεδο. Νομίζω ότι υπάρχει νομικό θέμα και υπάρχει και συνταγματικό θέμα. Αν δηλαδή αύριο ο πρόεδρος της Κένιας έρθει ε, στις development days και τον απειλήσετε με ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο δεν συνδέεται με το συνταγματικό χρονοδιάγραμμα που ορίζει, με το χρονοδιάγραμμα που ορίζει το σύνταγμα στη χώρα του. Τι κάνει κανείς, δεν παρεμβαίνει στα εσωτερικά ζητήματα της χώρας αυτής. Εσείς μιλήσατε για εκδημοκρατισμό των χωρών αυτών. Όλοι το ε, καλοδεχόμαστε, αλλά μήπως εμείς διακυβεύουμε αυτόν ακριβώς τον εκδημοκρατισμό. Γιατί υποσκάπτουμε ακριβώς αυτή τη νομική και συνταγματική κανονικότητα στις χώρες αυτές. Βεβαίω θα πρέπει να σκεφτούμε και ποιο είναι το πλαίσιο του ΠΟΕ μέσα στο οποίο εμείς μπορούμε να κινηθούμε. Μην ξεχνάτε πως ο κανονισμός πρόσβασης αγοράς για τις χώρες ΑΚΕ δεν ευθυγραμμιζόταν με τους κανόνους του ΠΟΕ. Αυτό ήταν ξεκάθαρο. Και θυμηθείτε πως μπορεί κανείς να λάβει εξαιρέσεις από τον κανονισμό του μάλλον ε, ε, κράτους εάν υπάρχει είτε ζώνη ελεύθερων συναλλαγών είτε ε, περιφερειακή συμφωνία. Οπότε προσπαθήσαμε να κάνουμε εμεί την περιφερειακή συμφωνία έτσι ώστε η προτίμηση που προσφέρουμε εμείς στις χώρες ΑΚΕ να ισχύσει. Και ο Ντέιβιτ και εγώ στην τελευταία θητεία δώσαμε μεγάλη μάχη για να δώσουμε περισσότερο χρόνο ε, και να δοθεί μια εξαίρεση από τον κανονισμό αυτό από τον ΠΟΕ. Οπότε η προθεσμία του Οκτωβρίου 2016 ήταν μια νίκη, μια επιτυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί πολλοί ζητούσαν να περιορίσουμε αυτή την προθεσμία. Υπάρχει λοιπόν το θεσμικό πλαίσιο για όλη αυτή την προσπάθεια. Δεν βασίζεται σε απόφαση απλώς Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Συμβουλίου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τώρα το λόγο για να απαντήσει και κυρίως για το θέμα ε, για τα θέματα κρέατος από ε, τον Καναδά, για παράδειγμα, και το κατά πόσο είναι αναπτυξιακή βοήθεια ή εμπόριο για τα χρήματα που θα χρειαστούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για το ε, παράδειγμα του τι έχουμε κάνει σε προηγούμενες συμφωνίες και όχι με τις χώρες Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους και ευχαριστώ πολύ για την ε, πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων σήμερα. Νομίζω πως έχουμε ακούσει το μήνυμα για την υπογραφή και έχω δει πολλούς υπουργούς και τον Ρομπ ε, Ντέιβις ανάμεσά τους πολύ ικανοποιημένους θεωρούν ότι διαπραγματεύτηκαν μία συμφωνία η οποία πρώτα απ' όλα είναι δίκαιη. Και αυτή τη λέξη τη χρησιμοποίησαν επανειλημμένα. Έπειτα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο σύστασης. Πιστεύω πως έχει περιγράψει πολύ σωστά τη συμφωνία και μάλιστα συμπεριέλαβε και μία ιστορική ανασκόπηση. Τώρα Νομίζω πως έχουμε την ευκαιρία να κλείσουμε, να ολοκληρώσουμε αυτό το έπος που άρχισε το 2000, όταν δηλαδή μετά τη συμφωνία του Κοτονού αναφερθήκαμε στις εμπορικέ συμφωνίες. Μετά λοιπόν από τόσα χρόνια και με τη συμμετοχή των χωρών και φτάσαμε σε αυτό το σημείο όπου υπάρχει αυτή η συμφωνία. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω τον κύριο Λάγκε, ο οποίος μας ανέφερε ότι έχουμε μια ιστορική ευκαιρία αυτή τη στιγμή και έθεσε τη συμφωνία και στα πλαίσια του ΠΟΕ. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικός ο έλεγχος που ανέφερε ο κύριος Σούστερ. Η παρακολούθηση. Ακούσαμε πολλές παρεμβάσεις και μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε κάποιες ιδέες. Θα σας ενημερώσουμε φυσικά. Φυσικά και υπάρχουν προϋποθέσεις μόνο εάν η εφαρμογή είναι σωστή, εάν συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών. Σίγουρα αυτά δεν θα τα αγνοήσουμε. Τώρα θα αναφερθώ στις ερωτήσεις σας. Να πω καταρχάς ότι και η Μποτσουάνα και η Βολιβία ε, βρίσκονται μπροστά στο, αλφάβητο στο λατινικό αλφάβητο, όμως πολύ πίσω οικονομικά σε, στην ανάπτυξη. Στην Μποτσουάνα δίνουμε μηδενικού, μηδενικές ποσοστώσεις, μηδενικούς δασμούς, αλλά όχι στην άλλη χώρα. Και μετά περνάμε σε αυτόν τον κανονισμό πρόσβαση στην αγορά. Καταρχάς, νομίζω πως είναι απίθανο να μην ε, κυρώσουν τη συμφωνία. Είναι δύσκολο βέβαια να φανταστεί κανείς ότι, μπορούν, ότι θα υπογράψουν ένα κείμενο που δεν έχουν διαβάσει. Πιστεύω πως το έχουν κάνει. Και πιστεύω πως μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Επίσης, κύριε Σόλτς, σωστά το είπατε, εμείς δεν θα εφαρμόσουμε προσωρινά την συμφωνία προτού αυτή επικυρωθεί. Πρώτα οι χώρες πρέπει να υπογράψουν και να επικυρώσουν τη συμφωνία. Δεν ζούμε στο 2008 όπου ενεργούσαμε βασισμένοι σε υπογραφές ή πολλές φορές μονογράφησης μιας συμφωνίας. Αυτό είναι κοροϊδία για τη δημοκρατία σε αυτές τις χώρες. Δεν αρκεί λοιπόν μία μονογραφή, μία υπογραφή και ε, εντάξει μετά είναι όλα καλά. Θυμηθείτε την περίπτωση της Βολιβίας. Πρέπει να γίνουν σεβαστές κάποιες προϋποθέσεις. Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι πάρα πολύ που αναφέρθηκε το πλαίσιο του ΠΟΕ. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι ως προς ε, την αντιμετώπιση των άλλων εταίρων. Τώρα, όσο και την ανάγκη να εξετάσουμε με περισσότερη λεπτομέρεια τις ε, διατάξεις. Όλες οι συμφωνίες το 2014 δεν έχουν την... Ε, δεν αναφέρουν να καταργηθούν οι, δασμ, οι δασμοί εξαγωγές. Τώρα, η ασφαλιστική δικλίδα για τις νεόφυτες βιομηχανίες. Το θέμα είναι τι εννοούμε με αυτόν τον όρο. Είναι τόσο ασαφείς οι ορισμοί που σε αυτές τις χώρες οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί νεόφυτο. Βρίσκονται ό, ε, όλες οι βιομηχανίες, οι επιχειρήσεις σε βρεφικό στάδιο, οπότε θέλει προσοχή. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, SPS χρειάζεται να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να καταργηθούν οι δασμοί. Θυμάμαι πολλούς ελεκτές οι οποίοι εξέταζαν ένα σώρο προϊόντα. Ναμίμπια, υδατοκαλλιέργεια για παράδειγμα. Υπάρχουν πολλά προϊόντα υδατοκαλλιέργειας από την Ναμίμπια που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή πληρούν τις προϋποθέσεις. Με την Μποτσουάνα τα προβλήματα που υπάρχουν είναι με ε, κάποια είδη βοηδών, με τα βουβάλια. Πρέπει να τους ε, βοηθήσουμε λοιπόν να βελτιώσουν ε, την παραγωγή τους περιφερειακά. Διότι διαφορετικά δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρουμε εδώ να γευτούμε αυτό το πολύ ωραίο κρέας βουβαλιού που δοκιμάσαμε στην Ποτσουάνα. Να σας υπενθυμίσω τώρα για τους ε, δίκαιους όρους ε, σε σχέση με τον ΠΟΕ. Δεν υπάρχει νομολογία ακόμα για αυτό το θέμα, όμως ε, το 80% είναι πολύ χαμηλό ποσοστό. Ελπίζω όλοι στον ΠΟΕ να κατανοήσουν ότι αυτό καλύπτει ένα ουσιαστικό μέρος του εμπορίου. Μετά, το θέμα δεν είναι τα ευαίσθητα προϊόντα, αλλά να έχουμε λογική στην αντιμετώπιση. Δεν πρέπει να υπάρχουν, ε, να υπάρχουν τρόποι να προσπεράσουμε την νομοθεσία. Στην περίπτωση της Μοζαμβίκης, για παράδειγμα, πιστεύω πως η διαφορά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ουσιαστική. Δεν ξέρω πώς μπορούμε δηλαδή να παρακάμψουμε την νομοθεσία και στην περίπτωση του dumping και πάλι και των επιδοτήσεων, εγώ θα έλεγα πως ε, τα προϊόντα μας είναι ανταγωνιστικά και ορισμένοι ε, έχουν ανάγκη αυτά τα προϊόντα, έχουν ανάγκη υψηλή ποιότητα τρόφιμα. Γι' αυτό λοιπόν το dumping δεν ανήκει στις πρακτικές μας. Τώρα, περιφερειακές συμφωνίες που μπλοκάρουν τις υπόλοιπες, ερώτησε η κυρία Σαρτζεντίνη. Ε, αυτό που συμβαίνει εδώ αντίθετα είναι, να, είναι ότι εμείς έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ καλό μέτρο σύγκρισης για παρόμοια προϊόντα. Και θα μπορούμε όλοι να υποφεληθούμε από αυτό. Οι κανόνες καταγωγής είναι πολύ σημαντικοί για όσες χώρες θέλουν να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία των προϊόντων τους. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη. Θέλουμε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στην Αφρική. Τώρα. Aid for Trade. Βοήθεια για εμπόριο. Πρέπει να καταλαβαίνόμαστε, να δούμε τι έχει γίνει. Θα έλεγα ότι ο Επίτροπος Λουί ε, Μισελ όταν ακόμα εργαζόταν στο χαρτοφυλάκιο των ε, συμφωνιών είχε ασχοληθεί και με τις περιφερειακές συμφωνίες. Δεν πρόκειται για τα ίδια κονδύλια. Το περιφερειακό χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαμβάνει και τη στήριξη του εμπορίου, ε, έχει κονδύλια ύψος 1,3 δις. Στα υπόλοιπα προγράμματα, περιφερειακά προγράμματα, το ποσό είναι 3,3 δις. Αυξήθηκε. Γι' αυτό λοιπόν δεν παρατηρείται σημαντική αύξηση, διότι η αύξηση αυτή είχε γίνει πιο πριν. Ίσως δεν ήταν ό,τι πιο έξυπνο κάναμε, όμως εμείς δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για την βοήθεια που δώσαμε. Και αυτό που κάναμε ήταν να φροντίσουμε πραγματικά να αποφεληθούν οι χώρες αυτές από την βοήθεια. Ελπίζω να κάλυψα όλα αυτά τα σημεία. Νομίζω οι συνάδελφοί μου δεν έχουν κάτι να προσθέσουν. Αλλά αν δεν κάλυψα κάτι, παρακαλώ, πείτε μου, Πρόεδρε. Ναι, ε, το κεφάλαιο σχετικά με την βιωσιμότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την μεταρρύθμιση Εδώ θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι. Όλα, όλες οι συμφωνίες συνδέονται με το κοτονού. Δεν υπάρχει δηλαδή μείωση των ε, προτύπων. Βιωσιμότητα. Τώρα, τι θέλουμε. Θέλουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε το πόσο συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών. Θέλουμε να συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών. Και από την εμπειρία μου έχω να πω ότι η κοινωνία των πολιτών έχει εργαστεί πολύ σκληρά για να συμμετέχει. Γι' αυτό θα ήθελα εδώ να έχω και την βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι είναι πολύ ε, σημαντικό να ε, μας βοηθήσετε για να γίνουμε πιο αξιόπιστοι εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΔΕΦΚΟ έχουμε δεσμευτεί για να συνεισφέρουμε οικονομικά στην βιώσιμη ανάπτυξη και στα διάφορα σχετικά έργα. Και σήμερα το απόγευμα όταν θα κάνουμε την ακρόαση για τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας θα ακούσετε περισσότερα. Ε, για μένα σημαντικό είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πρότυπα και προσπαθούμε να τηρήσουμε ε, τις ε, σχετικές ε, διατάξεις που έχουμε κατά της παιδικής εργασίας, κατά της ομοφιλοφοβίας. Γι' αυτό θέλουμε να υπάρχουν πραγματικές δομές παρακολούθησης έτσι ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε την εφαρμογή όλων αυτών των διατάξεων. Και να πω και ότι το έχει εκτιμήσει η κοινωνία των πολιτών αυτό, ότι εμείς τακτικά τους δίνουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν, να συνδιαλέγονται με τις κυβερνήσεις τους. Και πολλές φορές κάνει τη διαφορά μόνο ότι είμαστε εκεί. Γι' αυτό λοιπόν ε, σε καμία περίπτωση ε, δεν ε, μειώνουμε τις προδιαγραφές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ. Εργαλειοθήκη. Κανείς δεν ξέρει εάν είναι πλήρης. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό τα εργαλεία που υπάρχουν να χρησιμοποιούνται με το σωστό τρόπο. Ο εισηγητής έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, να μιλήσω για την περιαγωγή και την ενιαία αγορά. Πρώτη φορά ακούω αυτό το θέμα στην Επιτροπή Εμπορίου, όμως αυτή την ε, φορά δεν αναφέρεται στα κινητά, αλλά αναφέρεται στο κρέας ε, από βουβάλι. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ όλους για τα σχόλιά σας. Άκουσα πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις από τον κύριο Μάτα, τον κύριο Ζαραντήλ, τον Κρίστοφερ Φιέλνερ. Κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ σημαντικό ε, να γνωρίζουμε ότι η ημερομηνία είναι μια ημερομηνία που επιλέξαμε. Είναι μια επιτυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτή η ημερομηνία και ότι τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε ε, ακολουθώντας αυτό το χρονοδιάγραμμα. Δεν θα προσθέσω τώρα κάτι πάνω σε αυτά που είπε η Κομισιόν. Να πω όμως ότι ε, ο κύριος Σούστερ μας ανέφερε ότι υπήρχε έλλειψη ενθουσιασμού στις χώρες ΑΚΕ. Συναντήθηκαν όμως οι χώρες αυτές, αλλά και, καταλαβαίνω αυτήν την ε, έλλειψη ενθουσιασμού. Όμως σκεφτείτε και πόσες χώρες δεν ανήκουν στις χώρες ΑΚΕ, αλλά είναι αναπτυσσόμενες. Εδώ υπάρχει μια τεράστια διάκριση εις βάρον πολλών αναπτυσσόμενων χωρών και αυτό λόγω της ε, απικιοκρατικής μας ιστορίας. Τι κάνουμε δηλαδή, ακόμα βρισκόμαστε ε, σε αυτήν την θέση. Ζούμε μία μεταπικιοκρατική εποχή και έτσι αντιμετωπίζουμε τις χώρες εκεί. Και καταλαβαίνω λοιπόν την έλλειψη ενθουσιασμού για αυτές τις συμφωνίες. Όμως πολύ σωστά ο ΠΟΕ απεφάνθη ότι είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Τώρα, ο Κρίστοφερ νομίζω το παρατράβηξε μιλώντας για νέο υπεριαλισμό. Ε, εντάξει, είπε ψήγματα αλήθεια. όμως η αλήθεια είναι ότι αυτές οι χώρες υπέγραψαν μια συμφωνία. Και για μας θα ήταν αλαζονικό να τους πούμε ότι υπεγράψατε κάτι που δεν ξέρετε, δεν ξέρετε τι κάνετε. Και τέτοια σχόλια άκουσα σήμερα. Είναι κυρίαρχα κράτη αυτά. Κράτη με τα οποία διεξάγουμε συναλλαγές βασισμένα στη λογική και τα κράτη αυτά έχουν απόλυτη επίγνωση του τι κάνουν. Μόνο ένα με εξέπληξε. Αυτό που άκουσα, αν δεν κάνω λάθος, από την Μαρία, δεν θυμάμαι από ποιον, ότι, ότι οι ευρωβουλευτές δεν είναι ενημερωμένοι σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Δεν είναι δικό μας θέμα να ενημερώνουμε τους βουλευτές στην Αφρική. Είναι θέμα κοινοβουλίου αφρικανικού, αφρικανικής χώρας, των δικών τους πολιτικών ε, ανδρών. Ε, έχουν δέκα χρόνια στη διάθεσή τους για να ενημερωθούν. Νομίζω λοιπόν πως αυτή τη στιγμή φτάσαμε στη στιγμή να επικυρώσουμε τα όσα έχουμε συζητήσει. Και για το τελευταίο σημείο που είναι το monitoring, εδώ πιστεύω πως όντως μπορούν να γίνουν πολλά και μπορούμε να κάνουμε ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση αρκετά. Υπάρχουν αυτοί οι μηχανισμοί παρακολούθησης ε, οι οποίοι είναι μια πιθανότητα. Πρέπει να το κοιτάξουμε. Δεν έχω κάποια έτοιμη απάντηση, όμως μέχρι να έρθει η ώρα της επικύρωσης πρέπει να είμαστε επικοδομητικοί και να δούμε τι λειτουργεί και τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, έτσι ώστε στο τέλος να έχουμε ε, κάνει μια καλή δουλειά. Τώρα, ε, οι ρήτρε και τα άρθρα θα εφαρμοστούν και θα ισχύουν μόνο όταν ξέρουμε τι κάνουμε με το μηχανισμό παρακολούθησης. Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι πάρα πολύ που έχω την στήριξή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό η Μαρία. Ένα σύντομο σχόλιο μόνο. Να πούμε δηλαδή ότι επειδή τα κοινοβούλια υπέγραψαν όλα τελείωσαν, είναι σαν να λέμε ότι επειδή τα έχει υπογράψει ήδη η Κομισιόν και το Συμβούλιο, τι, γιατί να τα συζητάμε στο Κοινοβούλιο. Δεν συμφωνώ καθόλου. Έχουν υπογράψει και εμεί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα εξετάζουμε. Και το ίδιο ισχύει και για εκείνου. Ενώ το έχουν υπογράψει, παρόλα αυτά θα το συζητήσουν και στα Αφρικανικά Κοινοβούλια. Ακριβώ το ίδιο είναι. Και η συζήτηση πρέπει να γίνει όχι έτσι βιαστικά, αλλά με ένα εύλογο χρονικό διάστημα τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Εμεί αυτό λέμε, ότι πρέπει να υπάρξει ένα κοινοβουλευτικό διάλογο στην Αφρική. Γιατί μέχρι τον Οκτώβριο θα πρέπει να ακυρωθεί. Είναι σαν να του λέμε σε ένα μήνα πρέπει να ακυρώσετε την TTIP. Σαν να μα έλεγε κάποιο. Αλλιώ χάνετε τα πλεονεκτήματα. Όχι, δεν θα είμαστε ούτε εμεί ικανοποιημένοι ω ευρωβουλευτέ. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να σεβαστούμε τι αφρικανικέ δημοκρατίε. Για να σα απαντήσω εν συντομία, επί τη ουσία συμφωνώ πλήρω. Όμω δεν εναπόκειται σε εμά να δώσουμε τέτοιε συστάσει και οδηγίε στι αφρικανικέ χώρε ε, ω προ τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουν την κύρωση. Δικό τους ζήτημα είναι, εκτός μικροφώνου, τα σχόλια. Okay. Thanks a lot Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σόλτς, πολύ σύντομα. Επειδή αναφερθήκατε τώρα στο monitoring, συμφωνώ πλήρω, αλλά πριν περάσουμε στη φάση τη παρακολούθηση, πρέπει να ξέρετε ή να ξέρει κανεί το ακριβέ χρονοδιάγραμμα για τι ε, καταξιδότητε πράξει. Να απαντήσει σε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώ θα κινηθούμε ω προ αυτό. Η Κομισιόν. Χρονοδιάγραμμα για τι καταξιδότητε πράξει. Πολύ καλό ερώτημα. έχει ήδη αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση ουσιαστικά. Είχαμε την πρώτη συνεδρίαση στη διαδικασία των κατευθυντών συμπράξεων. Ουσιαστικά έτσι λοιπόν θα πάει στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο και τελικά το μπαλάκι θα πέσει στη δική σας μεριά. Σκλάβοι εμείς, αφεντικά εσείς. Εσείς θα μας πείτε τι θα κάνουμε. Καταληκτική προθεσμία 20 Ιουνίου για τροπολογίε και ψηφοφορία θα γίνει στις 13 ε, και 14 Ιουλίου. Εντάξει, ευχαριστώ. Ένα λεπτό διάλειμμα. Και μετά ξεκινούμε τη συνεδρίαση των συντονιστών και κλεισμένων των θυρών. Λίγοι μόνο επιτρέπεται να μείνουν.